Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε εδώ. Είναι μεγάλο προνόμιο για μένα να μιλώ σε εσά εδώ. Είναι δυναμική κοινωνία σήμερα και έχει μεγαλύτερες απαιτήσει για διασύνδεση ε, και ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε οι μεταφορές γίνονται ραχοκοκαλιά όσον αφορά την οικονομία μας και τις ζωές μας. Οι μεταφορές οθούν την ανάπτυξη και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμενοι για αυτή την ακρόαση παρατήρησα τυχαία ότι θεωρείται σαν δεδομένο ο τομέας των μεταφορών θεωρείται δεδομένος. Θα ήθελα να πω ότι υποτιμάται μάλιστα στην Ευρώπη σήμερα. Θεωρείται σαν πρόβλημα και όχι σαν μια λύση και όχι σαν δημιουργός θέσεων εργασίας. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να αλλάξω αυτή τη στάση συνεργαζόμενοι με εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να δώσουμε στις μεταφορές τη σημασία που τους αξίζει. Ήδη γνωρίζετε αυτή τη σημασία, το γνωρίζω, διότι ψηφίσατε να τριπλασιάσετε τη χρηματοδότηση για τις υποδομές για την τρέχουσα περίοδο του προπολογισμού. Έχω πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που μια τέτοια δέσμευση ε, μας ε, οδηγεί να αντιμετωπίσουμε και ελπίζω να αναγνωρίσετε σε μένα ότι με πάθος θα στηρίξω αυτό τον ζωτικό τομέα. Ξεκινώντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι οι μεταφορές πρέπει να είναι φιλικές στο περιβάλλον, πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τους πάντες. Διότι ας μην λησμονούμε ότι οι μεταφορές τελικά αφορούν τον κόσμο. Το κοινό που ταξιδεύει, τους εργαζομένους, εσάς και μένα. Όπως ο, ανάφερε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, το έργο της νέας του Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναπτυχθεί γύρω από την ανάγκη για δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την ανάπτυξη και να επικρατήσει τελικά η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας ε, κάθε στιγμή και θα πρέπει να εντάσσουμε αυτές τις αρχές σε κάθε πτυχή των μεταφορών και των συναφών πολιτικών. Ό,τι κάνουμε πρέπει να δημιουργεί αξία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Η πρώτερη επασχόλησή μου μου έδωσε πολλές εμπειρίες και ένα συνέστημα της σημασίας που έχουν τα δίκτυα. Όταν αναπτύσσουμε στρατηγικές με πελάτες και δήμους, η επιμελητία ήταν πάντα σημαντικό τμήμα αυτών όταν τα επεξεργαζόμαστε. Χρειάζεται σωστός εφοδιασμός, ομαλός και θα πρέπει να εντάσσεται το εφοδιασμό σε ένα ευρύτερο αποτελεσματικό δίκτυο. Και αυτό είναι το κλειδί στη σύγχρονη ζωή μα. Όπως γνωρίζει, όποιος έχει αναμειχθεί με την καινοτομία, ξέρουμε ότι γνωρίζει καλύτερα όταν υπάρχει υψηλή ποιότητα και λειτουργούσα υποδομή για να υποστηρίξει την καινοτομία. Στην περίπτωση των μεταφορών, οι υποδομές θα πρέπει να ενταχθούν σωστά και να είναι υποδομές συμβατές τεχνικά ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφορών που χρησιμοποιεί ο κόσμος, οδικές μεταφορές, υδρομικές μεταφορές, αερομεταφορές και ψηπλοεία. Επιπλέον υπάρχουν πολλές δυνατότητες για καινοτόμες ε, επιχειρήσεις και διάφορα σχετικά μοντέλα. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τη βέλτιστη διασύνδεση στην Ευρώπη ε, και θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα. Και γι' αυτό είναι κρίσιμο τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών να μετατραπούν σε πραγματικότητα θα πρέπει να κατασκευάσουμε τους κρίκους που λείπουν και θα πρέπει ε, τελικά να γίνει ομαλή κυκλοφορία. Είναι κάτι σημαντικό για αυτή τη διαδικασία. Υπόσχομαι ότι θα σημειώσω πρόοδο από αυτού. Υπόσχομαι επίσης ότι αν διοριστώ θα ηγηθώ των προσπαθειών για την εξέβρεση βέλτιστης της λύσης για ολοκληρωμένο σύστημα που θα λειτουργεί σωστά στην Ευρώπη, σύστημα μεταφορών. Εγώ είμαι μηχανικό και επιχειρηματία, Αυτό είναι το επαγγελματικό μου υπόβαθρο και βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε ε, πολλά με νέε τεχνολογίε για τι μεταφορέ, κυρίω με την τεχνολογία τη πληροφορική. Σεβόμενοι βέβαια ε, τις παραδοσιακές αξίες και τα πρότυπα τη Ευρώπη, κοινωνικά πρότυπα και περιβαλλοντικά. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά η πληροφορική μπορεί να είναι ένα έξοχο μέσο που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη επιτυχία. Θα ήθελα να αναφέρω απλώ μερικά από τα προγράμματα. Το e-call, το σύστημα πληροφορίας για την ποτάμευση πλοία και το σύστημα για τη μεταφορά μέσω σιδηροδρόμου, το ευρωπαϊκό σύστημα, το ERTMS. Τα δίκτυα των μεταφορών είναι και θα παραμείνουν βασικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης. Είναι η καρδιά της αλυσίδας εφοδιασμού που θα παρέχει ελεύθερες ροές αγαθών και ανθρώπων. Χρειάζεται διασύνδεση υψηλής ποιότητα σύγχρονες και λειτουργούσες υποδομές. Αυτά είναι ζωτικά για την ανάπτυξη. Αποτελούν ένα κομμάτι για την λύση όσον αφορά την ανάκαμψη της Ευρώπης, την οικονομική ανάκαμψη. Αν με εγκρίνει το Κοινοβούλιο σαν Ευρωπαία Επίτροπο, θα χρησιμοποιήσω την αποφασιστικότητά μου, την εμπειρία μου και την αφοσίωσή μου. Θα εξασφαλίσω ότι οι μεταφορές θα δώσουν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη και θα συμβάλλουν στην ε, στο πράσινο πρόγραμμα εφαρμογής μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πράσινο θεματολόγιο. Αστραφώ τώρα προς τις αρχές που θα αποτελέσουν κομβικό σημείο για τις προτεραιότητές μου για την επόμενη πενταετία. Θα ξεκινήσω επιστρέφουσα στη σημασία που έχει διαλειτουργικότητα και χρήση πολυτροπικών μεταφορών, διότι θα συμφωνείτε το μέλλον των μεταφορών είναι η διασύνδεση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε πολυτροπικό σχεδιασμό ταξιδιών, έκδοση εισιτηρίων, παρακολούθηση αγαθών, πραγματική προσμέτρηση του άνθρακα, διαθεσιμότητα και προστασία δεδομένων και αποδοχή αυτών. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα, θα πρέπει να έχουμε μια όθηση τεχνολογική που θα χρηματοδοτηθεί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι εμπλεκόμενοι φορεί του τομέα να συμμετάσχουν. Εάν τελικά με θα καλέσω όλους τους φορείς να καινοτομήσουν μεταφορές της πόλης, τις μεγάλες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέες εταιρείες, παρόχους δημοσίων μεταφορών και τα κράτη-μέλη. Οι πόλεις και αστικές περιοχές είναι καλός, καλό πεδίο δοκιμών για την καινοτομία. Πάρτε την πόλη μου, τη Λουμπλιάνα, πραγματο χάρη. Έχει πέντε λεωφορεία ευρυδική ε, κίνηση και είκοσι ε, λεωφορεία που κινούνται με μεθάνιο. Χάρη στο πρόγραμμα Σίβητα ε, τη Ευρώπη. Οι αρχέ τη πόλη προγραμματίζουν καθαρότερε, ασφαλέστερε και πιο αξιόπιστε δημόσιε μεταφορέ. Η πρωτοβουλία για τι ευφυεί πόλη, πιο συγκεκριμένα, έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σχετικά με αυτό, κυρίω για αυτό που συζητάμε θα είναι το πρόγραμμά μας ε, που θα ηγείται των προσπαθειών την επόμενη πενταετία. Θα πρέπει να τηρηθεί η ορμή του προγράμματος, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες όσον αφορά τις μεταφορές, την ενέργεια και τον τομέα ε, της πληροφορικής για να βελτιώσουμε το αστικό περιβάλλον της Ευρώπης. Θα ήθελα όμως επίσης να τονίσω ότι η πόλης, το smart cities δεν αφορά μόνο τεχνολογία αλλά και κοινωνική καινοτομία. Γι' αυτό η στενή συνεργασία πολλών εμπλεκομένων φορέων είναι κάτι που θα απαιτηθεί ούτως ώστε να αναγνωριστούν οι ευκαιρίες και να ακολουθηθεί η ορθή κατεύθυνση. Για το μέλλον τα ευφυή συστήματα μεταφορών, ITS, θα δραματίσουν σημαντικό ρόλο διότι εμπεριέχουν μεγάλο δυναμικό όσον αφορά την ασφάλεια, με οχήματα και υποδομές. Επιφέρουν και σημαντικά περιβαλλοντικά ωφέλη, διότι βοηθούν να αποφευθούν μη αναγκαίες διαδρομές και μετακίνηση κενών οχημάτων και μπορεί να είναι πιο αποδοτικό ο τομέας των μεταφορών και οι εκπομπές θα ελαχιστοποιηθούν. Και όπως έχει πει και ο πρόεδρος ο κ. Γιούγκερ αν η Ευρώπη θέλουμε να έχει φθηνή ενέργεια διαθέσιμη τα επόμενα χρόνια, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το μερίδιο των εναλλακτικών καυσίμων και ανανοσίμων πηγών ενέργειας στην ενέργεια που χρησιμοποιούμε. Οι μεταφορές έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε αυτή τη φιλοδοξία, διότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από το πετρέλαιο σαν πηγή ε, κινητήριας δύναμη. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι μεταφορέ έχουν ρόλο να παίξουν εξασφαλίζοντα ότι η Ευρώπη θα πετύχει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για την περικοπή των αερί, εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Εν αυτή την ενία θα εργαστώ για να συμβάλλω στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συντονίζεται και κατευθύνεται από τον Αντιπρόεδρο Σεφκοβίτς. Εναλλακτικά καύσιμα είναι στο επίκεντρο Τη ε, πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποια είναι η πρόκληση. Να ξεκινήσουν οι προσπάθειε και να λειτουργούν επιτόπου όλα αυτά τα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν επαρκείς υποδομές, ότι θα κατασκευαστούν αυτές, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ούτως ώστε αυτά τα καύσιμα να κινούν τον τομέα των μεταφορών στο μέλλον. Αλλά μη μην λησμονούμε και το σημαντικό ρόλο που θα παίξει και η τεχνολογία ούτως ώστε να στηριχθούν έτσι περαιτέρω αυτοί οι στόχοι. Αξιότιμα μέλη, ένα πράγμα το οποίο μάθαμε από το παρελθόν είναι ότι όταν δεν επενδύουμε σε μεταφορικές υποδομές διαπράττουμε ένα σφάλμα που έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε ότι οι μεταφορικές υπηρεσίες πάντα θα υπάρχουν για μας ή θα είναι πάντα ασφαλείς εάν δεν τις συντηρούμε τις υπηρεσίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι δημόσιες επενδύσεις ε, μειώνονται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Οι προπολογισμοί για συντήρηση και η ποιότητα των υποδομών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν μειωθεί. Θα πρέπει να δράσουμε και δεσμεύομαι να το κάνω αυτό. Επίσης θα κάνω ό,τι μπορώ ούτως ώστε να προωθήσω ολοκλήρωση μεταξύ διαφόρων μεταφορικών τομέων βάσει της αρχής των γενικών υποδομών και των κόστων που συνεπάγονται και θα χρηματοδοτούνται γενικές υποδομές από αυτούς που χρησιμοποιούν τις υποδομές. Αυτό θα γεννά εισόδημα και θα γίνει πιο πράσινο το σύστημα των μεταφορών. Χωρίς επενδύσεις κινδυνεύουμε να χάσουμε την ε, θέση μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό χρησιμοποιώντας καινοτόμα συστήματα χρηματοδότησης ούτω ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται προς βασικές υποδομές μπορούμε να δημιουργήσουμε, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα μια εποχή που η Ευρώπη τα χρειάζεται όλα αυτά πάρα πολύ. Η επένδυση των 300 δισεκατομμυρίων, το πρόγραμμα που πρότεινε ο πρόεδρος ο κ. Γιούνκερ, θα προσπαθήσει να καλύψει αυτή τη χρηματοδοτική ανάγκη δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης αμέσως και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον που θα το προστατεύουμε. Πρέπει να κάνουμε την καλύτερη χρήση των μέσων που διαθέτουμε. Πιστεύουμε ότι το μέσο για τη σύνδεση της Ευρώπης καθώς και τρόποι συμπλήρωσης εθνικών και περιφερειακών χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά Ταμεία και το Ταμείο Επενδύσεων είναι κάτι που χρειάζεται, αξιότιμα μέλη. Εάν ήθελα να συνοψίσω το ε, μελλοντικό μου θεματολόγιο, με μία λέξη θα έλεγα λαός, ο κόσμος. Πρέπει να έχουμε επίγνωση των κοινωνικών ζητημάτων και πώς επηρεάζονται από τις μεταφορές, πώς επηρεάζει τον τόπο εργασία ε, τομέα των μεταφορών, ε, τον τόπο εργασία, το εργατικό δυναμικό, την υγεία του, την ασφάλεια και την ισορροπία ιδιωτική ζωή και τόπο εργασία. Για εκείνου που εργάζονται το μεταφορικό τομέα πρέπει να επικρατούν κοινωνικέ συνθήκε δίκαιε. Ο μεταφορικό τομέα στο σύνολό του είναι γυράσκον τομέα, κυρίω όσον αφορά τι χεσέ μεταφορέ. Επιπλέον υπάρχουν σχετικά μικροί αριθμοί ε, γυναικών εργαζομένων σε αυτό το τομέα είναι σαφές ότι θέλουμε να αποφύγουμε στο μέλλον έλλειψη προσόντων παρά την υψηλή ανεργία που υπάρχει στους υπόλοιπους τομείς της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Οπότε θα πρέπει να γίνει ένα ελκυστικό επάγγελμα το μέσο των μεταφορών κυρίως για τους νέους. Θα κοιτάξω να δω ποια ευρωπαϊκή δράση μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να βελτιωθεί η κατάρτιση, να δημιουργηθούν προπτικέ για την απόκτηση προσόντων και να δώσουμε ποιοτικέ θέσει επασχόληση μεταφορέ. Πρέπει να υπάρχουν δίκαιε συνθήκες που επικρατούν. Και να το πω ξεκάθαρα, ε, είμαι κάθετα ενάντια στο κοινωνικό dumping. Η δικαιοσύνη όσον αφορά τι κοινωνικέ συνθήκε καθώ και τη εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι ουσιαστικά. Τέλο, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ενιαία αγορά. Είναι, μια... είναι ο στόχο Ευρωπαϊκή Ενώση, είναι η καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ενώσης. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα τη Ευρώπη για τι επιχειρήσει. Είναι ο κινητήρα που οδηγεί την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία, που βοηθά και τονώνει την σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι εξίσου ζωτική σημασία να αρθούν τα τελευταία τεχνικά και διοικητικά εμπόδια, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι μεταφορικές υπηρεσίες πραγματικά θα μπορούν να λειτουργούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί εθνικά όρια. Γι' αυτό προτίθεμαι να συνεργαστώ μαζί σας στενά και με το Συμβούλιο, ούτως ώστε να πετύχουμε την ταχεία έγκριση ε, του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και του τετάρτου πακέτου μέτρων για τους σιδηρόδρομους. Προέδρε, αξιότιμα μέλη, ίσως να βλέπετε στο άτομό μου ε, μία επίτροπο με ανοιχτό πνεύμα, υποψήφια επίτροπο, που έχει αφοσιωθεί, θα αφοσιωθεί μάλλον στην επίλυση των προβλημάτων με ένα καινοτόμο και συνεργάσιμο τρόπο. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για μας, το λαό και για να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Δεν μπορώ παρά να ελπίσω ότι αυτό βρίσκει απήχηση και σε εσά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμη να ακούσω τις ερωτήσεις σας.